θα ξεκινήσει αύριο το πρωί στις 9 μέχρι τη 1 και 3 με 7. Υπάρχει η η σε διάταξη που έχει δημοσιευθεί στο διαδίκτυο και λύγεται η συνεδρίαση. Ευχαριστώ.